έχουμε δύο κοινά πράγματα. Πρώτον, την ευθύνη μας απέναντι σε αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων. Άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν τις ελπίδες τους και τους φόβους τους. Και δεύτερον, όλοι είμαστε πολύ τυχεροί. Γιατί μια ζωή που την ξοδεύουμε στην υπηρεσία των άλλων είναι μια γεμάτη ζωή. Αλλά είναι γεμάτη μόνο εάν σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών των εκατομμυρίων ανθρώπων που είναι νοερά μαζί μας σήμερα εδώ. Εάν σκοντάψουμε, τότε οι πιο ευάλωτοι θα πληρώσουν το υψηλότερο τίμημα. Οι νέοι άντρες και γυναίκες που ψάχνουν το μέλλον τους και βλέπουν το κενό. Οι συγχυσμένε και παραζαλισμένε μητέρε πρόσφυγες, φύγοντα στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους, ξεσπιτωμένε, οι ανήσυχοι πατέρες, ανήμποροι να βρουν δουλειά για να θρέψουν του αγαπημένους τους. Και πολλούς άλλους που αισθάνονται στο περιθώριο, με την ταυτότητά τους να απειλείται. Το βασικό χαρακτηριστικό τη περασμένη δεκαετία είναι ότι οι άνθρωποι αποκτούν επιτέλου φωνή. Εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο ξεχύθηκαν στους δρόμους, έκαναν διαδηλώσεις, ε, καθιστικές διαμαρτυρίες, καταλήψεις, ε, ανέβασαν podcast και hashtag με τις επιθυμίες τους, ξεκάθαρα. Και όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα. Μια πραγματική ευκαιρία. Μια ευκαιρία να πολεμήσουν. Φίλοι, οι λαοί σε όλο τον κόσμο έχουν εκφράσει την θέλησή τους για το προορισμό που επιθυμούν. Αλλά θέλουν από εμά να τους καθοδηγήσουμε σε αυτήν την πορεία. Κοιτάν προς εμάς για να προβλέψουμε και να προετοιμάσουμε και να προλιάνουμε το έδαφος. Αυτό θέτει πολλά ερωτηματικά, πολλά και αν γίνει αυτό τι κάνουμε. Αυτές οι ερωτήσεις δεν είναι απλά καπρίτσια, δεν είναι ένα θεωρητικό εγχείρημα. Ειδικά στη δική μου περιοχή, όπου τα σενάρια τα χειρότερα βρίσκονται δυστυχώς πολύ κοντά στην πραγματικότητα και όχι στη σφαίρα της υπόθεσης και της εικασίας. Επιπλέον, αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τελικά τα αισθανόμαστε παντού σε όλο τον κόσμο, κατά κάποιον τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με τη βαθύτερη πληγή της περιοχής μου. Τι θα γίνει εάν ο κόσμος παρετηθεί από την λύση των δύο κρατών στη σύγκρουση Παλαιστινίων-Ισραηλινών. 70 χρόνια και πλέον πολέμου έχουν καταστρέψει τις ελπίδες για δικαιοσύνη. Σήμερα, αυτοί που είναι υπέρ της λύσης του ενός κράτους προσπαθούν να επιβάλλουν μια αδιανόητη λύση στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Ένα κράτος που θα στηρίζεται από θεσμικές ανισότητες με τους Παλαιστίνιους πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ένα κράτος που θα στρέφει την πλάτη στη γειτονία του, θα διαιωνίζει διαιρέσεις ανάμεσα στους λαούς και στις θρησκείες. Παγκοσμίω, πριν από πέντε χρόνια, ήμουν εδώ, σε αυτή την αίθουσα και μίλησα για τους κινδύνους του να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μην επιβάλλουμε την ειρήνη. Σήμερα θα πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι η κίνδυνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Υπάρχει βία ακόμη και περισσότερη. Αυξάνονται οι επικισμοί χωρίς να υπάρχει σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Το έχω πει άπειρες φορές, με διάφορους τρόπους και θα το ξαναπώ. Ξανά και ξανά. Ένας πιο ειρηνικός κόσμος δεν είναι εφικτός χωρίς μια σταθερή Μέση Ανατολή και μια σταθερή Μέση Ανατολή δεν είναι εφικτή χωρίς ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Τι θα συμβεί αν η Ιερουσαλήμ είναι μια, που είναι μια πόλη που την αγαπώ προσωπικά και έχει μεγάλη ιστορική σημασία για την οικογένειά μου, τι θα γίνει αν παραμείνει αμφισβητούμενη πόλη. Μπορούμε να στερήσουμε από τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους τις πνευματικές τους πεπιθήσεις, τα πνευματικά τους πιστεύω, την ειρήνη και την συνύπαρξη που συμβολίζει αυτή η πόλη και να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί πολιτική σύγκρουση. Ας ανεβάσουμε ταχύτητα και ας ε, σταθούμε λιγάκι στη διελκυστίνδα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι θα συμβεί εάν την επόμενη φορά καμία από τις δύο πλευρές δεν φύγει από την άκρη της Αβίσου και μας παρασύρουν όλους μας προς το χάος. Ένας ε, πόλεμος άνευ προηγουμένου μέχρι τα άκρα θα υποσκάψει τη σταθερότητα όλης της περιοχής, θα δημιουργήσει διαταραχές σε όλη την παγκόσμια οικονομία και στις ενεργειακές αγορές και θα προλιάνει το έδαφος για να δυθεί η τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τι θα γινόταν εάν, τι θα γίνει εάν το Ιράκ δεν καταφέρει να φτάσει στο ύψος των προσδοκιών ε, των πολιτών του, ε, να αξιοποιήσει το δυναμικό του και φτάσει πάλι σε έναν κύκλο 17 ε, ετών κλειδονισμών και ίσως ακόμα χειρότερα και ένοπλη σύγκρουση. Το Ιράκ είναι η χώρα με το 12% των παγκόσμιων πετρελαϊκών αποθεμάτων. Όμω, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι έχει 40 εκατομμύρια κατοίκου που έχουν υποφέρει μετά από τέσσερι δεκαετίε πολέμων, καταστροφικών κυρώσεων, κατοχή, ε, συγκρούσεων μεταξύ θρησκευτικών δογμάτων και του τρόμου του Άιζη. Σήμερα το μέλλον του ε, εναπόκειται σε μια ειρήνη πολύ ευάλωτη. Εγώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά δεν θα εγκαταλείψω τα αδέρφια μου εκεί. Τώρα, τι θα γίνει εάν η Συρία παραμείνει καθυλωμένη στις ε, παγκόσμιες αψημαχίες και ξεφύγει πάλι σε ένοπλο και εμφυλίο πόλεμο τι θα γίνει να αναδυθεί ξανά εκεί το ISIS και η Συρία γίνει το θέατρο επιθέσεων κατά του υπόλοιπου κόσμου. Η Συρία μπορεί να έχει βγει από τα πρωτοσέλιδα και από του πηχαίου τίτλου των εφημερίδων, και όμω ο πόνο δεν μπορεί να βγει από το μυαλό μα, διότι η κρίση δεν έχει περάσει. Τους τελευταίους μόλι εννέα μήνε, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν και πολλοί ήταν ήδη πρόσφυγες. Είναι κανείς εδώ σε αυτή την αίθουσα που θέλει να δει άλλη μια φορά κρίση προσφύγων από τη Συρία να ξεδιπλώνεται με όλη τη φρίκη και την οδύνη της. Θέλουμε να ξαναδούμε ένα αθώο παιδί να ξεβράζεται στις ακτές μας. Νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω την άποψη του καθενός και της κάθε μιας εδώ σήμερα, όταν λέω σε καμία περίπτωση. Και να σας ρωτήσω και το εξής. Τι θα γίνει αν καταρρεύσει η Λιβύη σε έναν πόλεμο άνευ ορίων και τελικά καταλήξει να είναι ένα κράτος αποτυχημένο. Τι θα γίνει αν η Λιβύη γίνει η Νέα Συρία, μια Λιβύη που είναι πολύ πιο κοντά στην Ήπειρο που είναι η πατρίδα μας. Ε, και να πω ξανά, τι θα γίνει αν αραβικές κυβερνήσεις... δεν καταφέρουν να δημιουργήσουν 60 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για τους νέους μας... τι ερχόμενες δεκαετίες. Και αν αποτύχουμε δεν θα δημιουργήσουμε τις τέλειες συνθήκες για την ανάδυση ε, ομάδων εξτρεμιστών. Η στρατολόγησή τους θα γίνει ακόμη πιο εύκολη εάν αφήσουμε πίσω μας ένα ίχνος ε, ευπάθειας και απελπισίας. Θέλουμε να αφήσουμε τους νέους αυτής της περιοχής να ζουν στην απελπισία και χωρίς ελπίδα. Φίλοι μου, αφήστε αυτόν τον στοχασμό με τις υποθέσεις του τι θα γινόταν εάν να γίνει μια επικοδομητική προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θα επιτρέψει να αποφύγουμε αναρρύθμιτες ε, τραγικές περιπτώσεις και να προστατεύσουμε τον κόσμο στην, στο ταξίδι του στη ζωή. Η πίστη μου στο Θεό ενισχύει την αισιοδοξία μου και την πεποίθησή μου ότι η ανθρωπότητα μπορεί να είναι δυνατή και ανθεκτική. Υπάρχει πάντοτε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ε, σε όποια μεριά και αν κοιτάξουμε, μια ε, εκδοχή όπου μας επιτρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η Αγία Γραφή, το Κοράνι, διδάσκει ότι αυτοί που μένουν καρτερικά και διατηρούν την πίστη τους στον Κύριο θα πάρουν τις μεγαλύτερες ανταμοιβέ. Η καρτερικότητα και η υπομονή είναι δύσκολες σε έναν κόσμο που δεν κατεβάζει ποτέ ταχύτητες, όπου σε κλάσματα δευτερολέπτου πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις και πρέπει να υπάρχουν αστραπιαία αποτελέσματα. Η η ηγεσία όμω, το να αναλαμβάνει κανείς ηγετικό ρόλο, απαιτεί το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή να μπορεί κανείς να στοχάζεται, να είναι σοφός και να έχει ένα μακρόπνο όραμα. Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε πολιτικούς με υπομονή και καρτερικότητα, διότι όλοι έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα των, ε, λαών μας και την ευημερία τους. Πρέπει να αντιδρούμε γρήγορα στα γεγονότα καθώς εξελίσσονται με ε, συγκρατημένες αποκρίσεις και όχι με σπασμωδικές αντιδράσεις. Η πολιτική δεν είναι ένα παιχνίδι που κερδίζει ο ταχύτερο. Καμιά φορά όσο ταχύτερα πηγαίνουμε τόσο πιο μακριά καταλήγουμε από τη γραμμή τερματισμού. Ο πατέρας μου, ο μακαρίτης ε, Βασιλεύς Χουσέιν, με είχε διδάξει ότι η ειρήνη είναι πάντοτε ο δυσκολότερος δρόμος, αλλά οδηγεί και στο υψηλό. Ένας δύσκολος δρόμος είναι ένας δρόμος που τον διαβαίνει κανείς καλύτερα με φίλους στο πλευρό του. Φίλους σαν εσά και τους λαούς της Ευρώπη, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα μέλλον όπου οι λαοί όλων μας ε, περιμένουν και που αξίζουν και εκείνοι και ολόκληρο ο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον ε, βασιλιά της ε, Ιορδανίας, έναν από τους ε, πιο σημαντικούς συνομιλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλο φίλο του Κοινοβουλίου και ακούσαμε τα λόγια του με προσοχή. Ευχαριστούμε για το πάθος και τον ενθουσιασμό για να επιδιώξουμε την ειρήνη, τον δημοκρατικό διάλογο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί. Και νομίζω ότι στις αρχές της φετινής χρονιάς βλέπουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη να δουλέψουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Δύο λεπτά και θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. και να president. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Επανάληψη της συνεδρίασης ε, και προχωράμε στις ψηφοφορίες. Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε μία ώρα και 20 λεπτά για τις ψηφοφορίες. Ε, με τη βοήθειά σας ε, ίσως να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Έχουμε πρώτα ε, την ε, πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Βισνιέσκα; Διαδικαστικό. Όχι, έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Συνάδελφε Κολάγια, σας παρακαλώ να ολοκληρώσουμε την ε, ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι? Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνάδελφε Κολάγια, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορούσατε να περιμένετε λίγο μέχρι να καθίσουμε όλοι ε, και να έχετε την προσοχή όλων, διότι πολύ θόρυβος γινόταν και δεν ακούγαμε τι λέγατε. Τώρα βέβαια ε, είναι πια αργά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά όμως, λέει ο Πρόεδρος. Ε, προχωράμε σε ψηφοφορία της έκθεσης Πορέμπα. Έναρξης ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Βαϊντέρε, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Φτάνουμε σε ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 45 ε, τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 46 ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, το αρχικό κείμενο ε, κατά τμήματα εγκρίνεται το πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση του τμήματος 2. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Το αρχικό κείμενο κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παραγραφος 3, αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολλές αποχές σε επαλήθευση. Ε, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία 47 υπέρ. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές πολλές αποχές επαλήθευση λοιπόν έναρξη της ψηφοφορίας ψήφισαν όλοι λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα και τα δύο με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, λήξη τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη τη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 28 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 49 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 σε δύο τμήματα, ονομαστικέ ψηφοφορίε και οι δύο, έναρξη τη ψηφοφορία για, την, για το πρώτο τμήμα. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 14. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, Έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, Έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 15. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση, έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι η λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παραχρός 16 σε 4 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Ζήτω συγγνώμη, λάθος μίλησα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Δύο φορές λάθος. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 58, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 73 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 22. Σε πέντε τμήματα αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι, λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Τροπολογία 1. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 23, αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα και τα δύο με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41 σε δύο τμήματα και τα δύο ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 24. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Ονομαστικές ψηφοφορίες. Σε πρώτο τμήμα έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 42 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 31 σε δύο τμήματα, ονομαστικές ψηφοφορίες. Πρώτο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, ονομαστική ψηφοφορία, της ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παραγράφος 27 σε δύο τμήματα. Δύο τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα, Έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλουμε επαλήθευση. Απορρίπτεται. 32 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 ονομαστική ψηφοφορία, ενάξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα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 Παραγράφος 34, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Κουραζόμαστε νομίζω. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 51. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 36. Επαλήθευση για την τροπολογία 51, έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 36, αρχικό κείμενο, τρία τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 72. Ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 70. Ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη τη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 40. Ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη τη ψηφοφορία.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 Έβδομο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 49, ε, αρχικό κείμενο, τέσσερα τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία για όλα, ε, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. η ψηφοφορία έρχεται αυτή. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Απορρίπτεται. 11 σε δύο τμήματα και ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πρώτο τμήμα. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο καταπίπτει. 54. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. 54. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 53 σε, 3, δύο τμήματα ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. χέρι. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 19 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. να απαντές πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία, ε, μάλλον εδάφιο 55, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται αυτή, ψήφισαν άπαντες. Πέρα. Εγκρίνεται. 7, τροπολογία 7, ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται αυτή. Εψήφισαν παντέ. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 αρχικό κείμενο στα τρία τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία για όλα. Πρώτο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. 57 αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται αυτή. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφο 60 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 61 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ Εγκρίνεται. 55, ε, τροπολογία 55, ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. ψήφισε ανάπαντε. Πέρας. Απορρίπτεται. 65 αρχικό κείμενο στα τρία τμήματα, όλε με ονομαστική κλίση. έρχεται αυτή. Ε, έρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Ψήφισε ανάπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56, ονομαστική ψηφοφορία. Ε, άρχεται αυτή. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 72 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο για την 72 δεύτερο τμήμα. Εψήφισαν άπαντε. πέρασε Εγκρίνεται. 73 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Εγκρίνεται. 34, τροπολογία 34, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75, αρχικό κείμενο. Εδάφη 75, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή να ψήφισαν Πέρας. Απορρίπτεται. 80 αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. 57 ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Έχουμε, το έχουμε κάνει αυτό. 83 αρχικό κείμενο. Σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. 35. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πέρασε 85. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59, ονομαστική κλίση, έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 36, ονομαστική κλίση, έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 ονομαστική κλίση αρκετή ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Ωραία. Έλεγχο για το τμήμα 2. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Επέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 90, αρχικό κείμενο, σε πέντε τμήματα, ονομαστική κλίση για όλα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα έρχεται η ψηφοφορία. Τέταρτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία και τώρα πε, λίγη εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίθηκε. 60 ονομαστική κλίση έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Απορρίπτεται. 91 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίν. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 64 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Εδάφιο 99, αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, κρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105, παράγραφος 105, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 62 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 13 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, πέρα. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο για την 107. Άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Εγκρίνεται. 63 τροπολογία 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Εγκρίνεται. 65 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Ε, ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Wir kommen nun zur Entschließung betreffend die Umsetzung und και τώρα θα περάσουμε στο ψήφισμα, στι προτάσει ψήφισμα του εφαρμογή παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στην Συμφωνία Αποχώρηση. Έχουμε έξι ε, με ονομαστική κλίση, παράγραφο 8, ε, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό τους, όπως δεν τροποποιήθηκε, έναρξη ψηφοφορίας, ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση της συναδέρφου ε, Βίζελερ Λίμα. Παράγραφος 3. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ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 Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ.